που θα έχει εγκρίνει και μελετήσει, ελέγξει μάλλον το φάκελο. Ναι, Επίσης, έχει εντελάβει το τελικό σχέδιο ημερησίας διάταξης ε, της 19ης Νοεμβρίου βάσει του άρθρου 137 του κανονισμού. Δεν υπήρξαν επίσημες αντιδράσεις, σχόλια, ούτε έτοιμα τροποποίησης του σχεδίου ημερήσιας διάταξης, οπότε θα θεωρήσουμε ότι αποφασίζεται έτσι η διάταξη των εργασιών μας. Όπως ε, προτείνει η διάσκεψη των Προέδρων στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι οι παρεμβάσεις διαρκείας.